στιγμή να απαντήσουμε στη Ρωσία. Υπάρχουν χιλιάδες πληροφορίες ε, που έχουν, έχει αποδειχθεί ότι ήταν ψευδής και θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει το δικό του ψήφισμα γι' αυτό. έχετε τον λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν για τη δήλωση. Να συνεχίσω τώρα τα εστονικά όμως. Η παραπληροφόρηση ε, δεν είναι κάτι καινούριο. Όμως κάθε φορά μας εκπλήσει όταν έχουμε ένα νέο κύμα παραπληροφόρησης. Είτε αυτό έχει να κάνει με τις ελεύθερες εκλογές, είτε έχει να κάνει με ε, επιθέσεις απέναντι σε κράτη-μέλη. Στα πλαίσια της κρίσης του κορονοϊού, αυτή η παραπληροφόρηση έφτασε σε νέα επίπεδα. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά τους λόγους που εμφανίστηκε ε, ε, ο κορονοϊός, ε, ψευδείς θεραπείες ε, και αυτά δεν έχουν τελειωμό και δεν θα τελειώσουν αν δεν κάνουμε κάτι. Πρέπει να αρχίσουμε να αντιδρούμε. Δεν είμαστε αρκετά αποφασιστικοί, δεν αντιδρούμε αρκετά γρήγορα. Ακόμα και σήμερα ακούμε αυτές τις δηλώσεις όπου μοιράζονται πληροφορίες που δεν βασίζονται σε δεδομένα ε, μιλάμε για συνεργασία με τις πλατφόρμες, το media. Πρέπει να λάβουν τις ευθύνες τους τα media. Και εμείς καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία της Κομισιόν για το θέμα της παραπληροφόρησης ε, ε, στα πλαίσια του κορονοϊού. Πρέπει να είναι τα δεδομένα ακριβή. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βασίζεται σε μια πρωτοβουλία κάποιων ανατολικών χωρών ε, δεν έχουμε την απαραίτητη εμπειρία ακόμα για να αντιμετωπίσουμε την προπληροφόρηση, αλλά πρέπει να δράσουμε και γρήγορα. Χρειαζόμαστε λοιπόν και χρήματα και, μέσα για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Πρέπει σε όλες τις χώρες της Ένωσης να κυκλοφορούν οι πληροφορίες σωστές και όχι μόνο σε κάποιες λίγες. Παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο σας, το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας, για να δείχνετε σεβασμό και στους συναδέρφους. Ο κύριο Κόρτσιτ. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ για τα βήματα που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τώρα, αλλά ε, κάπως προσεκτικά να τα δούμε. Θα λέγω ότι είναι ένα πρώτο βήμα σε ένα μεγάλο περίπατο που κάνουμε. Οπότε περιμένουμε νέες προτάσεις τους επόμενους μήνες. Τώρα, ε, σημασία έχουν λεπτομέρειες εδώ. Αυτή την βδομάδα φάνηκε ε, εμφανίστηκαν αποδείξεις δηλαδή για τις παρεμβολές της ε, Ρωσίας με παραπληροφόρηση μέσα στην Ευρώπη σε βάρος της Ευρώπης. Τι κάνουμε λοιπόν γι' αυτό. Αγαπητοί Επίτροποι, σκεφτείτε. Αν το κέντρο βάρους της δράσης αυτής το βάλαμε στις ε, κυρώσεις, αυτό θα τους εμπόδιζε να προωθούν και να δημιουργούν ιστοσελίδες και να πληρώνουν αυτούς που βρίσκονται πίσω από όλες αυτές τις δράσεις παραπληροφόρησης. <clears throat> θα κόστιζε δηλαδή στους αντιπάλους μας. Οπότε για να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον αυτή την παραπληροφόρηση αυτό πρέπει να κάνουμε. Συνεπώς, μην κοιτάμε μόνο και μην αναλύουμε μόνο τα συμπτώματα, αλλά και τις πραγματικές αιτίες που οδηγούν σε όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Λακαπέλ. Ο κύριος Λακαπέλ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελικά, δεν τρέπεται να μιλά για παραπληροφόρηση από πλευρά ιδιωτικών ή άλλων ξένων συμφερόντων στην πανδημία. Ένας εμπειρογνώμονας είναι ε, ο Μανουέλ Μακρόν. Είναι αυτός ο οποίος περιφρονεί την ομάδα μας όταν ζητήσαμε λόγω προφύλαξη να κλείσουν στις 24 Ιανουαρίου τα σύνορα. Η κυβέρνησή του μα απαντούσε όχι δεν έχει διαβατήριο ιό. Είναι αυτός ο οποίος για να κρύψει το γεγονό ότι δεν υπήρχαν μάσκε στη Γαλλία έλεγε ότι είναι περιττό να φοράμε μάσκες τι δράμα όμως αυτό όταν ξέρουμε ότι επειδή ακριβώς δεν υπήρχε προστατευτικό υλικό και εξοπλισμός έχασαν τη ζωή τους τόσοι γονείς και γιαγιάδες και παππούδες μας. Και υπουργό Υγεία που έλεγε ότι μαζική, μαζικός έλεγχος και εξετάσεις δεν ε, βοηθούν. Πάρα πολλά ψέματα λοιπόν από το ίδιο το κράτος που θα έπρεπε να είναι παραδειγματικό, με συνέπειες τραγικές και κάποιος θα πρέπει να λογοδοτήσει. Οπότε αγαπητοί εκπρόσωποι του Συμβουλίου και της Επιτροπής, μη μας δίνετε μαθήματα ηθικής για την παραπληροφόρηση όταν εσείς ήδη κάνετε ακριβώς αυτό. Ευχαριστούμε κυρία Βυσνιεύσκα. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Η παραπληροφόρηση αυτή δεν είναι κάτι καινούριο. Υπάρχει εδώ και καιρό. Τώρα όμως, χάρη στις νέες τεχνολογίες και σε νέες μεθόδους, η παραπληροφόρηση αυτή έχει καταστεί κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Σήμερα το συζητάμε και χτες το Κοινοβούλιο απέριψε την άρση ασυλίας ζητάει συγγνώμη γιατί δεν ε, μπορεί λέει, να προφέρει καλά το όνομα, ε, του κυρίου Φερχόφστατ. Και μάλιστα με έναν τρόπο ε, και τη στιγμή που το Κοινοβούλιο προσπαθεί να καταπολεμήσει την παραπληροφόρηση. Ενώ αυτά που είπε τη δείχνουν ότι τελικά μπορεί κανείς να λέει ψέματα στο Κοινοβούλιο, να σπείρει ε, μίσος να λέμε ότι είναι φασίστες τόσες χιλιάδες άνθρωποι όλοι αυτοί οι οποίοι διαδήλωσαν τον Μάρτιο 300 χιλιόμετρα στην Πολωνία από το Auschwitz. Όλα αυτά δείχνουν τελικά ότι το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί μια πηγή παραπληροφόρησης και διασπείρει ψευδείς ειδήσει. Αυτά και συγγνώμη. Όντως έληξε ο χρόνος είναι σημαντικό το θέμα βεβαίως, αλλά έχουμε περιορισμό χρόνου. Επόμενος, η κυρία Αντινόλφη. Παρακαλώ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι μάσκες έχουν σημασία μόνο για τους άρρωστους και τους υγειονομικούς. Οι μάσκες προστατεύουν τους άλλους. Υπάρχει μέσος κίνδυνος, υψηλός κίνδυνος, σοβαρή ασθένεια, καλό είναι να μην ταξιδεύετε και τα λοιπά. Ε, είναι σπάνιες οι περιπτώσεις ασυμπτωματικών, όχι τώρα παρακολουθούμε. Θα μπορούσα να συνεχίσω. Λοιπόν, πώς μπορούμε να μιλάμε εμείς για παραπληροφόρηση. Όλα αυτά τα έχει πει με την σειρά που τα ανέφερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ε, μιλάμε για οργανισμούς οι οποίοι υποτίθεται ότι ήταν έγκυροι, οι οποίοι έχουν πει τα πάντα και το αντίθετό τους ε, και βεβαίως ε, έχουμε αυτή την επίσημη υποτίθεται πληροφόρηση σε αντίθεση με το διαδίκτυο και από την άλλη είχαμε και τη δαιμονοποίηση της χώρας μου η οποία μάχεται και πολέμησε πρώτη στην Ευρώπη τον ιό. Λοιπόν, μία πρόταση είναι απλή. Να βοηθήσουμε τους πολίτες να έχουν τα εργαλεία ανάλυσης των πληροφοριών που λαμβάνουν, αλλά να προστατεύσουμε την ελευθερία έκφρασης. Θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα σταθερά τα οποία θα προωθούν τον μηντιακό αλφαβητισμό. Με συγχωρείτε λέει πρώτος, πρέπει να ολοκληρώσετε. Και ο επόμενος είναι ο κύριος Μπονιφέη. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είδαμε τους ε, μήνες αυτούς ε, μία συνεχή παραπληροφόρηση σε σχέση με το θέμα του κορονοϊού. Είδαμε να κυκλοφορούν ψευδείς ειδήσει κάθε είδους ε, και είχαμε τους Ευρωπαίους να στρέφονται ο ένας εναντίον του άλλου και να εξευτελίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα έχουμε μια ευκαιρία με το εγχείρημα αυτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ξεκινήσει μια ειδική επιτροπή που θα καταπολεμπά την παραπληροφόρηση και τις ψευδείς ειδήσει για να πολεμήσουμε αυτούς που θέλουν να διχάσουν τους Ευρωπαίους για συμφέροντα που είναι εξωτερικά. Το είδαμε αυτούς τους μήνες, αυτά τα χρόνια, ε, δημοσιογραφικές και δικαστικές έρευνες που αποκάλυψαν τη διαδρομή του χρήματος που στηρίζονται σε ένα λάθος δικαίωμα, δηλαδή την ενίσχυση επιπληρωμή της προπαγάνδας. Θέλουμε να υπερασπιστούμε την ελευθερία έκφρασης αλλά και να προστατευτούμε την δημοκρατία μας. Αυτό πρέπει να το κάνουν όλα τα θεσμικά όργανα. Σας ευχαριστώ. Τώρα όμως ζητώ συγγνώμη λέει η Πρόεδρος. Ξέχασα τον συνάδελφο Ανταμόβιτς. Βεβαίως έχετε δικαίωμα να μιλήσετε και πάλι συγγνώμη την κυρία Ανταμόβιτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι, σα ευχαριστώ. Να ευχαριστώ και την κυρία Γιούροβα για τι πληροφορίε που μα έδωσε, για την ενημέρωση, για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η καμπάνια παραπληροφόρηση είναι ένα μεγάλο κίνδυνο για τη δημοκρατία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κορονοϊό και η πανδημία μα το υπενθύμησε, υπενθύμησε αυτό ότι οι αξιόπιστε πληροφορίε μπορεί να σώσουν ζωέ. Το fake news, τα fake news όμως και το μίσος που, που διακινούν μπορούν να σκοτώσουν. Μπορεί κάποιο να κερδίσει την εξουσία, να μείνει στην εξουσία σε πολλά μέρη του κόσμου και στην Ευρωπαϊκή Ένωση χάρη στην παραπληροφόρηση. Ε, η δύναμη του ίντερνετ ε, έρχεται να διωγγώσει τη δύναμη της παραπληροφόρησης που κινείται πιο γρήγορα και από τον ίδιο τον ιό. Πρέπει να ε, βεβαίως να προωθήσουμε την ελευθερία λόγου. Όταν η ελευθερία λόγου χρησιμοποιείται για την παραπληροφόρηση, είναι το αντίθετο της ελευθερία. Οι που γίνονται με βάση μπλάθης πληροφορίες δεν μπορεί να είναι δημοκρατικές. Δεν μπορεί η ελευθερία να οδηγήσει, η υπερβολική ελευθερία να οδηγήσει την έλλειψη ελευθερίας τελικά άλλων. Πρέπει να μάθουμε, να διδάξουμε στους ανθρώπους πώς να, να, να αξιολογούν πληροφορίες. Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερο πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης και βεβαίως να υπάρχει πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία ο κύριος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, κύριε ε, Επίτροπε, κυρία Αντιπρόεδρε, το γνωρίζουμε ε, καλά ότι είναι καλύτερο να ακούει κανείς ε, ένα απλό ψέμα το οποίο να καθησυχάζει παρά μια πολυσύνθετη αλήθεια που ανησυχεί. Και αυτό συμβαίνει ακριβώς σήμερα. Ε, πάμε πολύ πιο γρήγορα με την παραπληροφόρηση και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε προφανώς. Το είπατε και οι δύο, το είπατε πολύ καλά. Είπατε κυρία Γιούροβα και το γνωρίζουμε όλοι προέρχεται από ένα καθεστώτα ολοκληρωτικά όπου η λογοκρισία ε, καθόριζε τη ζωή των ανθρώπων και δεν πρέπει να συμβεί αυτό για μα. Αυτό είναι το πρώτο λάθο που πρέπει να αποφύγουμε. Θέλω όμω να πιστώ την προσοχή σα και την προσοχή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε, σε ένα άλλο κίνδυνο που υπάρχει ε, δεν πρέπει να είμαστε αγαθοί. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ξένε δυνάμει που μα επιτίθενται. Γνωρίζουμε επίση ότι έχουν και διάβλου εντό των δημοκρατιών μα. Και οι φιλελεύθερε δημοκρατίε ε, ε, εκεί κινδυνεύουν. Ε, προσοχή λοιπόν, ούτε να πάμε προς τη λογοκρισία και να γίνουμε σαν τους ανταγωνιστές μας, ούτε όμως να εμπιστευόμαστε τυφλά την αγορά, διότι είδαμε ότι για την, τα ίδια στοιχεία παραπληροφόρησης η Google θα απαγορεύσει το Twitter όμως θα το αφήσει και θα τα εξηγεί και το Facebook δεν θα κάνει τίποτα στα πλαίσια της ελευθερίας της έκφρασης υποτιθέμενης. Δεν μπορούμε λοιπόν να ε, μπορούμε απλά να εμπιστευόμαστε τυφλά την αγορά, θα πρέπει να ρυθμίσουμε και εμείς και εμείς θα είμαστε το πλάι σας κύριε Αντιπρόεδρε και κύριε Επίτροπε. Ο κύριος Μάιερ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τίποτα δεν είναι απολύτως λάθο και τίποτα δεν είναι απολύτως σωστό, είχε πει ο Γκεν Ροτ. Και κάτι άλλο θα ήθελα να αναφέρω. Υπάρχει μια τεράστια περίπτωση παραπληροφόρησης. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί μιλάμε για την κυβέρνηση ενός κράτους μέλου. Μιλάω συγκεκριμένα για την αυστριακή κυβέρνηση όπου ο καγκελάριο στην αρχή τη κρίση αυτή σε ένα λόγο του είχε πει ότι προσεχώ όλοι θα ε, γνωρίζουμε όλους όσους πέθαναν από κορώνα. Κάτι το οποίο βεβαίως, ε, όλοι θα γνωρίζουμε κάποιον ο οποίος πέθανε από κορώνα. Ε, κάτι το οποίο βεβαίως δημιουργεί ανησυχία. Και βεβαίως ε, και ο Υπουργός ε, Υγείας είπε ότι έβγαλε ένα διάγραμμα διά, διάταγμα με το οποίο δεν επέτρεπε, τον κόσμο, δεν επέτρεπε στον κόσμο να συναντηθεί με τους οικείους του τις ε, διακοπές ε, του Πάσχα. Λοιπόν, θα πρέπει να δούμε τι έγινε με την μαζική πληροφορήση σε ένα κράτος μέλος. Σας ευχαριστώ και για ένα λεπτό. Κυρίες και κύριοι, η παραπληροφόρηση είναι ένα από τα πιο σκληρά μέτρα που έχουμε σε έναν ασύμετρο κόσμο. Ε, δημιουργεί πιέσεις, ε, καταλήγει σε χάος. Η παραπληροφόρηση ε, βασίζεται βέβαια στην έλλειψη διαφάνειας. Αυτό που είναι προβληματικό είναι το θέμα της δημοσιογραφίας και των κοινωνικών δικτύων. Σε αυτά τα δύο μέτωπα λοιπόν πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε τις σωστές πληροφορίες. Υπάρχουν πάρα πολλά ψέματα και μισές αλήθειες που κυκλοφορούν για την Πολωνία και την Ουγγαρία για παράδειγμα και ποτέ δεν διορθώθηκε αυτό. Επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Και αυτό είναι μια παραπληροφόρηση που υπάρχει με αρνητικές συνέπειες μάλιστα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την εικόνα της προς τα έξω. Οπότε να ελέγχουμε τα στοιχεία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για να καταπολεμήσουμε την παραπληροφόρηση. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι πρέπει να περιορίσουμε το διαδίκτυο. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σταλέχος, ευχαριστώ πολύ. Μία από τι συνέπειε τη διαδικτυακή επανάσταση είναι ο ρόλο των μέσων ενημέρωση που φιλτράρουν την πληροφορία κανονικά την ενημέρωση γιατί φροντίζουν να κυκλοφορεί μόνο εκείνη η ποιότητα τώρα πια δεν μπορούν να το κάνουν αυτό και αυτό είναι ένα κενό το οποίο με κάποιο τρόπο πρέπει να καλύψουμε και γι' αυτό πρέπει να δούμε τι ευθύνη μπορούν να έχουν οι πλατφόρμες με την τεχνολογία που υπάρχουμε σήμερα και με κάθε προσοχή βέβαια ε, μπορούμε έτσι μέσω αυτών να βοηθήσουμε την ε, αποφυγή της παραπληροφόρησης. Να δούμε λοιπόν τι ρόλο παίζουν και τι ρόλο παίζουμε και εμείς όλοι οι χρήστες. Ας κοιτάξουμε τι γίνεται σε εμά, γιατί ε, βέβαια οι κυβερνήσεις πρώτα απ' όλα πρέπει να δεσμευτούν για διαφάνεια στις πληροφορίες που δίνουν και να φροντίσουν να είναι αξιόπιστες και πραγματικές να μην ακούμε περίεργα πράγματα και υπερβολικά, για παράδειγμα, για το τι μπορεί να κάνει η χλωρίνη και πώς μπορεί να βοηθήσει την καταπολέμηση του κορονοϊού. Να προσέξουμε λοιπόν τι κυκλοφορεί, όλα αυτά φυσικά και είναι παραπληροφόρηση επίσης. Η κυρία Μπάσο έχει τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ. έχουμε εδώ πέρα μια έλλειψη πυθούς. Λέτε ότι δεν θέλετε να περιορίσετε την ελευθερία έκφρασης, αλλά ταυτόχρονα θέλετε να μπλοκάρετε τους λογαριασμούς εκείνους οι οποίοι διαδίδουν ψευδείς ειδήσει. Να υπενθυμίσω εδώ πέρα ότι οι επαγγελματίες της ενημέρωσης συχνά είναι απλώς όργανα προπαγάνδας. Θυμόμαστε ότι στην Ιταλία στήριξαν την θέση της κυβέρνησης που ε, γνωρίζουμε πόσα, ε, πώς κατέληξε όσον αφορά το COVID. Όσον αφορά λοιπόν το θέμα του COVID, θέλετε απλά να βάλετε φήμοτρο σε όσους λένε άβολες αλήθειες. Λοιπόν, οι ψευδείς ειδήσει καταπολεμούνται με την αλήθεια, όχι με τη λογοκρισία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα περνάμε στην κυρία Σόφκο. Κυρία Πρόεδρε, για πάνω από τέσσερις ε, μήνες ε, αντιμετωπίζουμε μια πανδημία άνευ προηγουμένου η οποία έχει αλλάξει τις ζωές μας δραματικά και μας έχει αναγκαστεί, αναγκαστεί να προσέχουμε Καταφέραμε να παραμείνουμε ενωμένοι όμως και με αλληλεγγύη. Όμως η πανδημία αυτή δεν είναι η μόνη μάχη που δίνουμε βλέπουμε ένα τεράστιο κύμα παραπληροφόρησης για τον κορονοϊό που στόχο έχει να μας παρουσιάσει ως αναποτελεσματικούς και διχασμένους. Η εκστρατεία αυτή είναι ιδιαίτερως διαδεδομένη στα Δυτικά Βαλκάνια όπου στόχο έχει την αποσταθεροποίηση της περιοχής και να στρέψει την κοινή γνώμη ε, μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε στήριξη άνευ προηγουμένου 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά τη διάρκεια της κρίσης. Και όμως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι περισσότεροι πολίτες θεωρούν ότι άλλες δυνάμεις παρήχαν περισσότερα. Ο καλύτερος τρόπος είναι με διαφάνεια, λογοδοσία και μεγαλύτερη επικοινωνία. Γι' αυτό καλωσορίζω τις προσπάθειες της Stratcom και του συστήματος ε, ταχείας αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά και εμείς ως εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών. Πρέπει να κάνουμε το βήμα πάρπερα. Οπότε, περνάμε τώρα στην ολοκλήρωση της συζήτησης. Αυτή την φορά τον λόγο έχει η κυρία Γιούροβα να μιλήσει πρώτα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και σίγουρα δεν είναι η τελευταία φορά που συζητάμε για την δύναμη που έχει το διαδίκτυο και σωστά, γιατί βλέπουμε τη δύναμη αυτή καθημερινά. Βλέπουμε ότι το διαδίκτυο αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για να βοηθήσουμε με ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά μπορεί επίσης να είναι και ο χώρος όπου από την άλλη μεριά λαμβάνουν χώρα διάφορες παραβιάσεις, πραγματικές παραβιάσεις. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα λοιπόν για να το συζητήσουμε. Μόλις ξεκινήσαμε όπως είπα και πριν. Έχουμε το πρόγραμμα δράσης της Ευρώπης για το θέμα αυτό ε, μπροστά μας. Θα δούμε πώς θα προστατεύουμε τις εκλογές, για παράδειγμα, από την παραπληροφόρηση και από την εξωτερική ανάμειξη. Ε, θα δούμε το θέμα της δημόσιας συζήτησης, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται για να πουληθούν προϊόντα, αλλά χρησιμοποιούνται επίσης για να πουλήσουν και τους πολιτικούς ή τις απόψεις τους. Είναι ένα νέο στοιχείο λοιπόν στην πολιτική συζήτηση. Είναι κάτι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις εκλογές. Όλα αυτά τα θέματα που είναι ουσιαστικά πρέπει να τα συζητήσουμε και είναι και πολύ λεπτά. Οπότε, Περιμένω τη συζήτηση και τις συζητήσεις μάλλον που θα ακολουθήσουν και ελπίζω ότι μέχρι τα τέλη της χρονιάς θα είμαστε σε θέση να δούμε πώς ε, προχωράμε ε, στην ε, ανακοίνωσή μας γιατί υπάρχει εκεί κατάλογος με πράγματα που θα πρέπει να γίνουν μέχρι τότε και ελπίζω να έχουν πράγματι προχωρήσει και να δούμε και τι κοινέ λύσεις μπορούμε να βρούμε μεταξύ μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Αντιπρόεδρος, ο κύριος Μπορέλ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση που ε, σίγουρα δεν κλείνει το ζήτημα. Είχαμε σημαντικές συνεισφορές, ενδιαφέρουσες, ε, κάποια εξαιρετικά πρωτότυπα όπως ε, το να πούμε ότι η παραπληροφόρηση έχει τη ρίζα του στον Αδάμ και στην Εύα. Δεν ήξερα ότι ο Αδάμ ήταν ε, θύμα της παραπληροφόρησης από την Εύα ε, που δεν τον ε, ειδοποίησε για τις επιπτώσεις του να φάει το μήλο. Μπορεί, μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Εν πάση περιπτώσει, στον δικό μας κόσμο, τον τωρινό, πρέπει να αναγνωρίσουμε κάτι το οποίο είναι στη βάση και της όλης συζήτησης. Η δημοκρατία είναι ένα σύστημα που λειτουργεί με βάση την πληροφορία που έχουν οι πολίτες στη διάθεσή τους. Οι, οι, πολίτες επιλέγουν, εκλέγουν και για να το κάνουν αυτό πρέπει να γνωρίζουν ποιες είναι οι επιλογές που έχουν, πρέπει να αξιολογήσουν τη δράση των κυβερνήσεων και γι' αυτό χρειάζεται ελευθερία πληροφόρησης, πλουραλισμό και χρειάζεται και ακρίβεια στην πληροφόρηση αυτή. Εάν λάβουν λαθασμένες πληροφορίες οι πολίτες, δεν μπορούν να κάνουν και σωστές επιλογές. Είναι σαν ένα αεροπλάνο το, το οποίο το σύστημα πλοήγησης είναι χαλασμένο. Κάποια στιγμή θα πέσει. Είναι λοιπόν σημαντικό να δώσουμε αυτή τη μάχη έτσι ώστε πληροφορίες, η πληροφορία γενικά που θεωρούμε ότι είναι δημόσιο αγαθό να είναι στη διάθεση των πολιτών και να μπορούν οι πολίτες να επαληθεύσουν κατά κάποιο, κατά πάσο ε, κάποιος ε, τους κοροϊδεύει κάποιος τους λέει ψέματα. Ό,τι και να λέει ο αστριακός ποιητής που αναφέρατε, εγώ δεν νομίζω ότι πάντα υπάρχει ένα μέρος αλήθειας και ένα μέρος ψέμα, ε, μη αλήθειας στα πάντα. Κάποια πράγματα είναι σίγουρα αληθινά και κάποια πράγματα είναι σίγουρα ψέματα. Το ότι δύο ε, συν δύο μας κάνει τέσσερα στο δεκαδικό σύστημα ε, είναι αλήθεια, 100%. Κάποια πράγματα επίσης είναι εντελώς αναλυθεί όπως και αν το λέει. Το να υπάρχουν βεβαίως στοιχεία υποκειμενικά, ε, μπορεί κάποιος να έχει επιχειρηματολογεί υπέρ ή κατά του ενός ή του άλλου ζητήματος λόγω της ιδεολογίας του, προφανώς. Αλλιώς δεν θα είχαμε και πολιτική συζήτηση. Ένα πράγμα όμως είναι να αξιολογεί κάποιο υποκειμενικά τα δεδομένα και άλλο πράγμα είναι τα ίδια τα δεδομένα. Και όπως είπε η συνάδελφο, εμείς δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα, το Υπουργείο Αλήθειας. Είχε Υπουργείο Αλήθειας στην ε, χώρα του, είχα και εγώ στη χώρα μου, στην Ισπανία, όταν υπήρχε Υπουργείο πληροφορία. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε λοιπόν ένα Υπουργείο που θα ελέγχει το τι γνωρίζουμε και τι όχι. Θέλουμε να βοηθήσουμε τους πολίτες να μπορούν οι ίδιοι να διακρίνουν την αλήθεια από το ψέμα. Και, αυτό, και αυτή είναι η βάση ενό δημοκρατικού συστήματο. Ιδάλω ε, η δημοκρατία μα ε, θα είναι εντελώ ατελή και στο τέλο δεν θα είναι καν δημοκρατία. Ε, γι' αυτό χρειαζόμαστε υποστήριξη των δημοκρατικών δυνάμεων όλου του κοινοβουλευτικού τόξου έτσι ώστε να μπορέσει να επιβιώσει η δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε και ακούμε και την κυρία Υφυπουργό, την κυρία Νάτης. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρίες και κύριοι βουλευτές. Το θέμα αυτό είναι θέμα προτεραιότητας για εμάς. Πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες μας από την παραπληροφορία σεβόμενη την ελευθερία του λόγου και των μιμή. Οι κοινέ αξίες μας και τα δημοκρατικά θεσμικά άργανα έχουν μεγάλη σημασία για να μπορέσουν να ανταποκριθούν ε, στις ε, προκλήσεις. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε οριζόντια, διασυνοριακά και διακλατικά για να ανταλλάξουμε ευελιστές πρακτικές. Αναμένουμε την συνεργασία με εσά, με την Κομισιόν, την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση για να καταπολεμήσουμε την επιδημία παραπληροφόρησης. Οι πρωτοβουλίε αυτές όπως το σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία ή ο νόμος περί ψηφιακών υπηρεσιών θα μας δώσουν τη δυνατότητα να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση για αυτό το θέμα της ημερησιάς διάταξης ε, και περνάμε στην κοινή συζήτηση για την σύντομη παρουσίαση της έκθεσης Αουστρεβίτσιους, σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς Συμβούλιο Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής για θέματα ανατολικής εταιρικής σχέσης. Τον λόγο έχει ο κ. Πικούλα. Να σας υπενθυμίσω και πάλι ότι δεν θα έχουμε μπλε κάρτες και και οπότε έχουμε μια πιο σύντομη συζήτηση. Τον λόγο έχει λοιπόν ο κύριος Αυστρεβίτσιος. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, είπατε εκπρόσωπε. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω του σκιώδει εισηγητέ και όλου του βουλευτέ που συνεισέφεραν στην έκθεση αυτή. Πρόκειται για στενότερε σχέσει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έξι χώρε εταίρου. Πρόκειται για θετικά ε, βέβαια βήματα που γίνονται για την γειτονία μας, κάτι το, από το οποίο θα εξαρτηθεί ο ηγετικό ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απαιτεί ισχυρή δέσμευση. Μια τέτοια δέσμευση πρέπει να αποδειχτεί μέσω ενός μηνύματος ιστορικά αποδεδεγμένου προς τους εταίρους μας. Ότι δηλαδή αναγνωρίζουμε τις προσπαθειές σας και με συνεργασία μεταξύ μας θα σας βοηθήσουμε για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Είναι θέμα χρόνου. Το μότο μας για τις επόμενες ε, δεκαετίες της ε, ανατολικής γειτονίας θα πρέπει να είναι περισσότερα για περισσότερα και σταδιακά να υπάρχει ενσωμάτωση ε, σιγά σιγά ανάλογα με τα αποτελέσματα και βάση αρχών. Λυπάμαι που φεύγει ο κύριος Μπορέλ, αν και βλέπω τον Επιτρόπο Βαρέλη εδώ, αλλά μετά θα αναφερθώ σε αυτόν. Στον πολιτικό χώρο πάντως οι εταίροι μας θέλουν να συνεχίσει η στήριξή μας και να τους βοηθήσουμε με οδηγίες για την ενέσχεση της δημοκρατίας του κράτους δικαίου και την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Οικονομικά θα πρέπει να επιτρέψουμε την πρόσβαση στην ενιαία αγορά δημιουργώντας έναν κοινό οικονομικό χώρο. Μην ξεχνάμε ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι ενιαία δεν μπορούμε να στρέφουμε το βλέμμα μόνο στην ανατολική ή τη δυτική διάσταση. Μία υπάρχει, ευρωπαϊκή, και τώρα πρέπει να δράσουμε για αυτήν. Κυρία Πρόεδρε, η τη δυτικη διασταση μια υπαρχει η ευρωπαικη και τωρα πρεπει να δρασουμε γι αυτην κυρια προεδρε η πρωτοβουλια για την ε, ανατολική σχέση είναι μια επιτυχία και θα παραμείνει επιτυχία όσο συνεχίζουμε να δρούμε μαζί, από κοινού, με κοινό όραμα και κοινέ δράσεις, διάλογο και εταιρική σχέση. Κύριε Επίτροπε, όπως ε, γνωρίζετε από τα σημερινά νέα από την Προεδρία της Λευκορωσίας, ο επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος εκεί πέρα έκοψε τις πλευρές ως διαμαρτυρία για τα όσα συμβαίνουν. Θα ήθελα την αντίδρασή σας παρακαλώ. Είναι θέμα ανθρωπισμού αυτό. Ακολουθεί ο κύριος Πίκουλα. madam president Ευχαριστώ. Θα μιλήσω σήμερα για το μέλλον της ε, διεύρυνσης. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω τους σκιώδεις ε, εισηγητές ε, για την αφουσίωσή τους στην κοινή μας προσπάθεια. Το βασικό μήνυμα εδώ πέρα είναι να δώσουμε στήριξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η διεύρυνση είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο που έχουμε στην εξωτερική πολιτική για να επεκτείνουμε τις ε, αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, τον σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου. Η έκθεση αυτή τονίζει κάτι το οποίο συχνά ξεχνάμε η προοπτική ένταξη για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και προς το συμφέρον των χωρών που θέλουν να ενταχθούν. Για πρώτη φορά μετά από την ένταξη της Κροατίας το 2013 έχουμε και πάλι πολιτική ένταξης. Καλωσορίζουμε λοιπόν την θέληση του, ε, και την έγκριση του Συμβουλίου για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία. Θα πρέπει τώρα να δοθεί μια ημερομηνία. Θα θέλαμε να δούμε τα κεφάλαια να κλείνουν με γρήγορο ρυθμό και να υπάρξει μια πιο αποτελεσματική παρακολούθηση της ε, πρόοδου τους. Βεβαίως αυτό απαιτεί και τον ε, κατάλληλο προϋπολογισμό. Όσον αφορά τον ρόλο του Κοινοβουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να ενδύνει την στήριξη της ένταξης των Βαλκανικών χωρών. Τέλος, η διεύρυνση είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε να είμαστε αξιόπιστοι μόνο αν είμαστε βεβαίως ε, και πιστευτοί στην άμεση γειτονία μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξ ονόματος της ε, Επιτροπής, ο κύριος Επίτροπος, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες ε, και κύριοι βουλευτές, για την γεωπολιτική μας επιτροπή. Η επαφή με τους γείτονές μας έχει πρώτη προτεραιότητα. Αυτά δεν είναι μόνο λόγια, πρέπει να γίνουν και πράξεις. Να ξεκινήσω με τα Δυτικά Βαλκάνια. Τους πρώτους έξι μήνες της ε, θητείας μας είχαμε μια νέα μεθοδολογία για να γίνουν διαπραγματεύσεις πιο αξιόπιστες, ε, πιο δυναμικές ε, και με ισχυρότερη πολιτική κατέθεση. Και παρά την πανδημία, τον Μάρτιο το Συμβούλιο ενέκρινε μία απόφαση για να ξεκινήσουν εντεξιακές διαπραγματεύσεις με Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία και χαίρομαι για το ότι επιβεβαιώθηκαν αυτές οι αποφάσεις από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να στηρίξουμε την περιοχή αυτή κατά τη διάρκεια της πανδημίας ε, δώσαμε 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία κινητοποίησαμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Επιπλέον είχαμε και ένα αριθμό πρωτοβουλειών που κανονικά ισχύουν μόνο για τα κράτη-μέλη. Τον Δε Μάιο είχαμε την σύνοδο του Ζάγκρεμπο που οι ηγέτες ε, βεβαίω επέδειξαν την αλληλεγγύη τους ε, με την περιοχή και έστειλαν ένα μήνυμα ενισχυμένης ε, εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανατέθηκε στην Κομισιόν να καταρτήσει ένα σχέδιο επενδύσεων για την επιτάχυνση αυτών και των μεταρρυθμίσεων. Αυτή την εβδομάδα η Κομισιόν θα προτείνει το σχέδιο πλαισίου διαπραγματεύσεων ε, προς το Συμβούλιο, καθώς και μια ενημέρωση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Αναμένουμε την συνέχεια. Η διεύρυνση ε, είναι αξιοκρατική και για να υπάρξει μια πρόοδος. Οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων θα πρέπει να συνεχίσουν τι μεταρρυθμίσει. Απαιτείται περαιτέρω εργασία στα θέματα κράτου δικαίου, καταπολέμηση διαφθορά και οργανωμένου εγκλήματο, καθώ επίση και σε ζητήματα θεμελιωδών και ανθρωπινών δικαιωμάτων. Απτέ μεταρρυθμίσει σημαίνει να προχωράμε πιο γρήγορα στι συνταξιακέ διαπραγματεύσει. Και βεβαίως ε, το φθινόπωρο ε, θα καταρτήσουμε και ένα σχέδιο για να στηρίξουμε την οικονομική ανάκαμψη και να έρθει η περιοχή αυτή πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σχέδιο αντικατοπτρίζει πολλούς τομείς ε, που ορίζει η έκθεση σας, όπως η συνδεσιμότητα, ειδικά στον τομέα των μεταφορών και της ενέργειας, πράσινη μετάβαση και ψηφιακό μετασχηματισμό. Το σχέδιο αυτό θα φέρει ανάπτυξη και δουλειές στην περιοχή επίσης ως ε, τμήμα των κοινών προσπαθειών μας για την ανάκαμψη μετά την πανδημία. Τώρα, να εστιάσω στην Ανατολική γειτονία. Να σας ευχαριστήσω για την στήριξή σας ε, στην πολιτική μας. Η δέσμευσή μας ε, ως προς την Ανατολική γειτονία τονίστηκε και στο τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών. Είμαι πεπισμένος ότι θα επαναβεωθεί και στην συνάντηση των ηγετών αργότερα σήμερα. Στόχος μας είναι να οικοδομήσουμε με τις χώρες εταίρους ε, μια φιλόδοξη εταιρική σχέση που θα ε, συνεχίσει να έχει απτά αποτελέσματα για τους λαούς της περιοχής. Χαίρομαι λοιπόν για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει σχεδόν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ στις χώρες αυτές ε, μετά τον COVID-19. Έτσι έχουμε Ε, την ε, στήριξη αυτή για τις άμεσες χρηματοδοτικές τους ανάγκες και την ενίσχυση της μακροοικονομικής σταθερότητας. Έτσι θα, σωθούν και οι θέσεις εργασίας ε, με την παροχή ρευστότητα σε ολόκληρη την οικονομία και άμεση στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τονίζεται έτσι πόσο σημαντική είναι η ανθεκτικότητα ως συνολικό πλαίσιο των σχέσεών μας που θα είναι στο επίκεντρο του σχεδίου μας. Έχουμε λοιπόν πέντε στόχους πολιτικής. Πρώτα απ' όλα να εργαστούμε προς ανθεκτικές οικονομίες. Δεύτερον, να στηρίξουμε την ανάπτυξη θεσμικών οργάνων λογοδοσίας, κράτους δικαίου και ασφάλειας. Τρίτον, να στηρίξουμε τον πράσινο μετασχηματισμό και την κλιματική αντοχή. Τέταρτον, να στηρίξουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό και πέμπτον, να εργαστούμε προς την ανάπτυξη ανθεκτικών και δίκαιων συμπεριληπτικών κοινωνιών. Μαζί λοιπόν με τα κράτη-μέλη, χώρες εταίρους και άλλους θα διαμορφώσουμε τα παραδοτέα του 2020 που θα εγκριθούν στη Σύνοδο του Βερολίνου. Βασιζόμαστε λοιπόν στην ε, στήριξή σας ε, για να υπάρχει εταιρική σχέση τα επόμενα χρόνια. Και τέλος, προς τον ε, εισηγητή θα εξετάσω το ζήτημα το οποίο αναφέρατε. Τώρα το άκουσα, δεν το γνώριζα. Και βεβαίω θα ένα λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η κοινή συζήτηση. Αύριο η ψηφοφορία για την πρώτη έκθεση, για την έκθεση Πιτσούλα αύριο, οπότε η συνεδρίαση θα διακοπεί στις 11.45 και θα επαναληφθεί το φόβο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Δεν νομίζω πια άλλο. AUTHORWAVE